Ε, έβαλα γέρο στην κάρτα μου, αλλά έχω υπερψηφίσει το ψήφισμα. Το σημειώνουμε. Ευχαριστώ. Έχω λάβει λοιπόν την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Κυρία Έρκ, παρακαλώ. Δεν δούλεψε το μηχάνημά σας για την ψηφοφορία. Το σημειώνω. Άλλος, προχωρώ λοιπόν στα πρακτικά της συνεδρίασης θα συμπεριληφθούν όλα αυτά που σας έλεγα. Έχουμε τρεις μήνες ε, προθεσμία αρχής γενομένης ε, της αυριανής ημέρας 10 Σεπτεμβρίου του 2010. Τώρα, στη συνεδρίαση της 11 Νοεμβρίου του 2009, το Ευρωπαϊκό